Παρακαλώ καθίστε. Επαναλαμβάνεται η περίοδος συνόδου που διακόψει 26 Νοεμβρίου. Τα συνοπτικά πρακτικά και τα κείμενα που εγκρίθηκαν στις 26 Νοεμβρίου διατίθενται. Έχετε αντιρρήσεις, ενστάσεις από αυτόν. Όχι. Εσείς κύριε Γκέρικε θέλετε το λόγο παρακαλώ. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, σήμερα η μερίσια διάταξη έχει 7 συζητήσεις και 3 ψηφοφορίες και τίποτα δεν είναι επίγον. Παρακαλώ ε, από ε, το Προεδρείο να ελέγξει την πολύ ε, ακριβή όσο και άχρηστη σύνοδο στις Βρυξέλλες. Τι δουλειά έχει αυτό με τα πρακτικά κύριε Γκέρικη που λέτε, παρόλα αυτά θα εγγραφούν στα πρακτικά. Για τα πρακτικά λέγαμε τις προηγούμενες συνεδρίασης. Έχετε καμιά αντίρρηση, καμιά παρατήρηση, εγκρίνονται. και κύριοι, οι αρμόδιες πολωνικές αρχές με ενημέρωσαν για την εκλογή των κυρίων Χότς και Κλωρόσοβσκι από 27 Νοεμβρίου 2015 και έρχονται να αντικαταστήσουν τον κύριο Κρόβατσικ και τον κύριο Γιατσικίεβιτς καλωσορίζω τους νέους συναδέλφους και σύμφωνα με τον κανονισμό μας έχουν πλήρη δικαιώματα.